στο διάστημα τριών μηνών από τώρα. Στο επόμενο σημείο είναι συζήτηση για, τα, για τις παραδιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων δημοκρατίας και του κράτους δικαίου μία ώρα.